σε διάφορες γλώσσες εκ μέρου ε, τη ομάδα ID, Ταυτότητα και Δημοκρατία, κυρίως η κυρία Μπενιό. Συνάδελφοι, η COP15 τον Οκτώβριο θα πρέπει να θέσει στόχους για τα μελλοντικά χρόνια σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις διαδικασίε που έχουν προκαλέσει οι κλιματικές αλλαγές και κυρίω οι ανθρωπογενείς. Όμως είναι σαφές ότι συνεχώς να κάνουμε κηρύγματα στους πολίτες και να επιβάλλουμε και άλλους φόρους δεν είναι μάλλον η καταλληλότερη πολιτική ε, λύση. Ούτε η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, ούτε η αμφισβήτηση των συμφωνίων ελεύθερων συνεργών, ούτε η ανάγκη θέσπιση εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντο. Βεβαίω είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο διαβίωσή μα και του τρόπου κατανάλωση. Χρειάζονται προσωπικέ προσπάθειε φυσικά, αλλά δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα εάν δεν ε, υπάρξει ρήξη με τι ιδεολογικά δόγματα που μα επιβάλλονται. Πρέπει αμέσω να προστατεύσουμε τα είδη που απειλώνται από τι κλιματικέ και περιβαλλοντικέ αλλαγέ. Η κατάσταση στου πόλου και στην Αυστραλία μα το θυμίζουν με τρόπο δραματικό. Η υγεία των συμπατριωτών μα από την ατμοσφαιρική ρήπανση, τη ρήπανση των υδάτων, τη ρήπανση των εδαφών, από την λογική του κέρδου και τα οικονομικά συμφέροντα απειλούνται. Γιατί όμω να την πληρώνει ο ε, πολίτη που έχει ανάγκη το αυτοκίνητό του για να πάει να δουλέψει, ενώ οι θαλάσσιε μεταφορέ ή οδικέ μεταφορέ να μην αντιλαμβάνουν καμία υποχρέωση να μειώσουν του ρήπου του. Εδώ λοιπόν και λόγω των όσων ψηφίζονται τώρα ε, μπορεί να εξάγουμε με μεγάλα έξοδα ε, προϊόντα κακή ποιότητα στην άλλη άκρη του κόσμου ή να περνάμε νομοθεσία για τον περιορισμό τη χρήση ε, φυτοφαρμάκων και γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών και όλα αυτά ενώ μα προσφέρονται στο πιάτο άλλα που είναι εξίσου επικίνδυνα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ελεύθερη έκφραση και για την ε, και κάνουμε τα ανάποδα από αυτά που διακηρύσουμε στις εξαγωγές μας. Δεν πρέπει να είναι απλώς ωραία λόγια η οικολογία. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές αυτά, πραγματικά αυτά προβλήματα της εποχής μας. Ε, και τώρα, εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Βόντρα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η προστασία της βιοπικιλότητας είναι θέμα καθοριστικό, κρίσιμο και είναι πολύ επίκαιρη η συζήτησή μας γιατί σήμερα κιόλας το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημοσίευσε έκθεση για την ε, δραματική κατάσταση της βιοπικιλότητας και τις απώλειές της ανά τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πράγματα δεν εντοπίζονται τόσο πολύ στην Ευρώπη αλλά εκτός τα χαρτιά, τα κείμενα που ετοιμάζουμε εδώ στο κτίριο αυτό, πέραν κάποιων σημαντικών συστάσεων και μέτρων, όπως το να προστατεύσουμε τα, ε, τα, τους οικοτόπους, τα ενδιαιτήματα, το πώς να σταματήσει η αποψήλωση των δασών, πολλές φορές συγχέονται και με σοσιαλιστικά μέτρα που θέλουν να δώσουν μια άλλη κατεύθυνση στα πράγματα. Εν τέλει δεν θα είναι τόσο χρήσιμα όλα αυτά και θα φέρουν ε, τα αντίστροφα αποτελέσματα, πιστεύω. Εν είδη παραδείγματος για τα μεγάλα σαρκοφάγα, λιοντάρι, τίγρη και λύκο. Τα είδη αυτά ζουν σε χώρες επανάπτυκτες έχουν προβλήματα. Ενώ ο λύκος που ζει σε χώρες σύγχρονες όπως η Ευρώπη δεν απειλείται. Ίσα ίσα έχει αυξηθεί ο πληθυσμός ε, των λύκων. Έχει πολλαπλασιαστεί. Τα βήματα λοιπόν που ε, θα κάνουμε θα πρέπει να μην φέρουν ε, αρνητικά αποτελέσματα αλλά θετικά. Ευχαριστούμε συνάδελφε και τώρα από την Γκουε ο κύριος Μόντιγκ. Ευχαριστώ πολύ. Η βιοπικιλότητα είναι σημαντική αξία από μόνη της. Ε, έχει να κάνει όμως και με το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Όσο μεγαλύτερη βιοπικιλότητα, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να μετριάσουμε την αλλαγή του κλίματος. Πρόκειται για επίγον θέμα. Καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα η ε, βιοπικιλότητα και γι' αυτό είναι λυπηρό και απίστευτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε στην επίτευξη των στόχων για το 2020. Ε, θα πρέπει όμως πρώτα να αναστρέψουμε την τάση και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τις αιτίες. Αιτίες είναι η γεωργία, ο τρόπος διαχείρισης των δασών, ε, καθώς και η αλλαγή χρήσης γης. Θα πρέπει να πετύχουμε και τους στόχους του Παρισιού και τους στόχους ε, βιοπικιλότητας. Αυτή τη στιγμή δεν τους πετυχαίνουμε. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από γεωργικές πρακτικές όπως είναι οι μονοκαλλιέργειες και η διαχείριση των δασών είναι σημαντική διότι το 80% των ειδών στην Ευρώπη ζουν στα δάση. Η χρήση των δασών είναι πολύ σημαντική λοιπόν. Μιλάμε για αποψήλωση των δασών Ε, το πρόβλημα είναι όμως ότι μία φορά εξαφανίζονται τα είδη και πολύ μεγάλος αριθμός ειδών απειλείται. Για το έτος 2030 ε, χρειαζόμαστε αριθμητικούς στόχους και θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το 30% της βιοπικιλότητας. ευχαριστώ, Εύη. 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα δείχνει ξεκάθαρα τη δραματική κατεπίγουσα κατάσταση που ζούμε σε οικολογικό επίπεδο. Είναι μπροστά στα μάτια όλων μας ότι η καταστροφή της, φύ, φύσης είναι άνευ προηγουμένου ε, για πρώτη φορά. Ε, που επαπειλούνται ε, μιλάμε για ένα επιπλέον εκατομμύριο ε, νέα είδη που βρίσκονται σε, στον κίνδυνο της ε, Οι τρομερές ε, κλιματικές αλλαγές ε, κάνουν πολύ πιο δηλητηριώδη την απώλεια της βιβλιοποικιλότητας. Αυτή η τάση έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο το ανθρώπινο είδος και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο 80% των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Προβλήματα σε, στην ανθρώπινη υγεία, στην ε, διατροφική ασφάλεια κλπ. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει η τρέχουσα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη COP15 στην Κίνα είναι να προωθήσει την νέα στρατηγική για την επικοινότητα για το 2000 και να ξεπεράσει τη λογική των εθελοντικών δεσμεύσεων να έχει πιο φιλόδοξους στόχους, νομικά δεσμευτικούς για τη βιοποικιλότητα και την, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο σας και τώρα ο κύριος Λίζε για ένα λεπτό. Δεν τον βλέπω εδώ. Επομένως, Μπορεί αν ξαναμπεί στην αίθουσα να του δώσω το λόγο μετά. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Γκούτελαντ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εξαφάνιση ειδών ε, ε, γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι ε, παλαιότερα και αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική ε, οικολογική κρίση. Ένα εκατομμύριο ήδη, απίστευτος αριθμός, ε, απειλείται από εξαφάνιση. θυμόμαστε την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, αλλά η απώλεια βιοπικιλότητας θα έχει καταστροφικές συνέπειες για εμά του ανθρώπους. Εάν εξαφανιστούν ε, οι μέλισσε, τι θα γίνει ε, με την παραγωγή τροφίμων στον πλανήτη μας. Ε, ταυτόχρονα βλέπουμε συνέχιση χρήσης φυτοφαρμάκων στην γεωργία και γνωρίζουμε ότι είναι μία από τις αιτίες της κρίσης που ζούμε. Θα πρέπει να μειώσουμε τις ποσότητες χημικών στο περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι η ε, χρήση αυτή είναι επικίνδυνη. Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι ε, ουσίες που προκαλούν ορμονικές διαταραχές είναι επικίνδυνες και για το οικοσύστημα και για εμάς, τους ανθρώπους. Είναι όμως κάτι που υπάρχει στην καθημερινότητά μας και τα παιδιά μας ε, το ζουν αυτό στην καθημερινή τους ζωή. Είναι κάτι που απειλεί και τη δική μας υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για τα φυτοφάρμακα. Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που έχει γίνει και οι προτεραιότητες της πολιτικής μας ομάδας ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ψήφισμα για την COP15. Χαίρομαι που έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τη βιοπικιλότητα. Θα αγωνιστούμε για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, συνάδελφε. Σας συγχαίρω και για το όμορφο μωράκι σας που, μας, που σας συνόδευσε σε αυτή την παρέμβαση. Καμφά για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Επίτροπε, καλησπέρα. Συζητάμε σήμερα το βράδυ τη στρατηγική σας για τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη για το, μέχρι το 2030. Πολύ ωραία. Υπάρχει όμως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 και απέτυχε πλήρως. Κανένας από τους στόχους προστασίας της φύσης στην Ευρώπη που είχαμε θέσει δεν υλοποιήθηκε. Αν έρθετε προς εμάς τέλος Φεβρουαρίου, σε λίγες εβδομάδες, με μια στρατηγική, με μεγάλα νούμερα, με ωραίες προθέσεις, αλλά τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα νομοθετικό, τίποτα δεσμευτικό που θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε τα δεδομένα, τότε θα είναι μια συμπαθητική στρατηγική, ομορφούλα, αλλά περιττή. Αυτό που περιμένουμε συγκεκριμένα είναι 30% του συνόλου της ευρωπαϊκής επικράτειας να προστατεύεται για να αφήσουμε λίγο ήσυχη τη φύση κατά της ε, επίθεσης και των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θέλουμε στόχους μείωσης συγκεκριμένων με νούμερα ε, για τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη. Τι επιθυμούμε. Να έρθετε επιτέλους με μία μέθοδο προστασίας και αξιολόγησης επίπτωσης αυτών των φυτοφαρμάκων στις μέλη σας. Εδώ και μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας έβαλε Σα έθεσε το ερώτημα. Περιμένουμε ακόμα τη νέα σα πρόταση. Και επίση πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση εκτό Ευρώπη. Εμεί, η Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είμαστε αυτή που επηρεάζει περισσότερο με την κατανάλωσή τη τα τροπικά δάση. Α επανέλθετε με μια συγκεκριμένη πρόταση κατά πολέμηση τη αποψήλωση εκεί. Αυτό θέλουμε. Εάν δεν τα έχουμε αυτά, κύριε Επίτροπε, τότε θα είναι μια στρατηγική κενή περιεχομένου. Ευχαριστώ. Και τώρα, Τουσά. Ένα λεπτό, κυρία Τουσά. 75% του χερσαίου εδάφου και 65% του θαλάσσιου εδάφου ε, απειλούνται. Ένα στα 8 είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό καταστρεφόμαστε. Το μέλλον της ανθρωπότητας απειλείται από αυτές τις ε, επιθέσεις που ε, με πολυεθνικές οι οποίες ε, καταστρέφουν τα δάση, ε, καταστρέφουμε τη φύση για να ρέει το πετρέλαιο. Εδώ και πολύ καιρό ε, το χρήμα πριν τα ανέβει στα σύνορα θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις εθνικές στρατηγικές και λογικές αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα κοινό μας αγαθό. Αντί να επιθέμεθα στη φύση και να την εκμεταλλευόμαστε χωρί ήκτο, θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ω ένα πλανητικό κοινό που έχει το δικαίωμα να νεωθεί. Εδώ δεν πρόκειται για φιλοσοφικές συζητήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει νομική κακό καθεστώ στη φύση για να προστατεύσουμε ό,τι ζει. Την επόμενη χρονιά ε, είναι πολύ σημαντική για αυτό. Ε, ο ΙΕ ζήτησε ε, συγκεκριμένους στόχους. Αν δεν θέλουμε να αποτύχει η COP15 ή όπως η COP25 θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καταστρέφουμε και σκοτώνουμε τη φύση. Και το δικαίωμα στη φύση που έχει η φύση στη ζωή. Ευχαριστώ. Λίμερ για δύο λεφτά. Συνάδελφοι, ποιος από εμά ε, δεν θέλει καθαρό αέρα, καθαρά ποτάμια ε, και προστασία ε, της χλωρίδας και της πανίδας. Συμφωνώ μαζί σας με λογικό τρόπο να εργαστούμε πάνω στις συνθήκες πλαισίου. Ε, μας περιμένουν πολύ έντονες συζητήσεις. Για μένα ο άνθρωπος είναι μέρος του οικοσυστήματος. Ε, αλλά ε, πολύ εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χωρίς ε, τους ανθρώπους όλα θα ήταν καλύτερα. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει σταυροφορία για, για τον μετριασμό του κλίματος. Αλλά βλέπουμε πώς υπέφτουν θύματα αιωλικών πάρκων στην περιοχή τους με ψέματα. Ε, υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν ε, στην ε, καλύτερη πιστοποίηση προϊόντων. Εγώ γελάω όμως με όλα αυτά. Ε, κάποιοι ε, ε, βρίσκουν λυπηρή την εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών. Άλλοι αναφέρονται στις πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου της υπεράκτιες. Άλλοι μιλούν για τα φυτοφάρμακα ενώ πολλοί από αυτούς ε, δεν ασχολούνται καθόλου με τα επικίνδυνα χημικά στις μπαταρίες ε, στην ε, Κίνα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η αλλαγή του βιολογικού περιβάλλοντος είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Αν λοιπόν ε, συνεχιστεί αυτή η ρητορική, ε, τότε μάλλον ε, σε λάθος αιτίες Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Υπάρχει, συνάδελφοι, υπάρχει γαλάζια καρδιά. Σας τη δέχεστε. Συνάδελφε Λίμερ, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε. Από τον συνάδελφο Μέτς. Με συγχωρείτε, αλλά αρνήθηκε συνάδελφος. Και τώρα ο κύριος Μπομπάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η τελευταία έκθεση τη Διαπαιδευτική Πλατφόρμα για την Βιβλιοποικιλότητα μα ανησυχεί πάρα πολύ. Πάνω από ένα εκατομμύριο ζωικά είδη και φυτικά είδη, ένα στα οκτώ δηλαδή, απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι η έκτη μαζική εξαφάνιση που λαμβάνει η χώρα στον πλανήτη. Και όμω δεν έχουμε λάβει τι σωστέ αποφάσει. Ούτε καν του στόχου του 2010 δεν έχουμε επιτύχει. Οι αποφάσει λοιπόν τη COP15 θα είναι κρίσιμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δραστικά μέτρα και το ίδιο και η διεθνή κοινότητα. Εγώ προτείνω ήδη δύο. Πρώτα απ' όλα για τα φυτοφάρμακα. Βάσει των επιστημόνων, η εντατική ε, γεωργία είναι ένα βασικό λόγο απώλεια τη βιοπικιλότητα. Τα φυτοφάρμακα όπω ο γλυφοσάτη, ε, μεγάλη ευρύτατη χρήση, είναι υπεύθυνα για πολλά από αυτά τα φαινόμενα. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει για την απαγόρευση με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προβλέποντα συγκεκριμένε εναλλακτικέ. Επίση, η γάμα τα χρησιμοποιούνται για την ε, ε, διατήρηση τι καλλιέργειε με αυτοφάρμακα. Το 2001 είχαμε ήδη τότε απαγορεύσει τι τεχνικέ, όμω οι μεγάλε εταιρείε προσπαθούν να παρακάμψουν τι νομοθεσίε τα νομοθετικά μα μέτρα, με ε, την ε, εισαγωγή άλλων γάματα φόμικρων που καταστρέφουν το περιβάλλον μα. Και πρέπει και πάλι να αναλάβουμε δράση για να είναι κατάφοροι κατά δίκη του και η απαγόρευσή του. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κ. Μάμερη για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Μάμερη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επερχόμενη Σύνοδος για την Ποικιλότητα θέλει να δημιουργήσει μέτρα για το μέλλον όλων των ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμεί δεν κοιτάμε εδώ την συμπεριφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρει μόνο να παίρνει και να ξαναπαίρνει και να παίρνει κι άλλα. Δείτε στα βρετανικά ύδατα πόσα είδη ε, ε, χάνουν τη ζωή του λόγω των Ιλλανδικών αλληλευτικών ε, ε, σκαφών που χρησιμοποιούν ε, ηλεκτροσόκ για τα ηλεκτρικά μέτρα ή για τα τεράστια αλλιευτικά σκάφη που σαρώνουν ολόκληρα κοπάδια ψαριών και ό,τι άλλο βρεθεί στο διάβα τους ε, και μαζί και πολλές φορές τα έξυπνα και κοντινά στον άνθρωπο δελφίνια. Αυτά τα αλλιευτικά, τα τράτες καταστρέφουν τα είδη και έξω από και στα νυχτά χωρών της Αφρικής και καταστρέφουν ένα σωρό είδη. Είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το προβάδισμα στο κέρδο και όχι στη βιοπικιλότητα. Πρέπει να πάψουν οι πρακτικέ που απειλούν το περιβάλλον ε, ήδη εδώ. Ε, στη δική μας την αυλή δεν μπορούμε να δίνουμε, να, κάνουμε, να φωνούμε κηρύγματα κατά τον άλλον. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Λίνς για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η βιοπικιλότητα και η προστασία του κλίματος πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είχαμε φιλόδοξους στόχους στη Σύνοδο των Παρισίων ε, προηγουμένως, αλλά τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο και στη βιοπικιλότητα. Χρειαζόμαστε ένα ηχηρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας κοινότητας. Θα πρέπει να συνδυαστούν η προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομία και να υπάρξει μια συνεισφορά για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Έχουμε τη δυνατότητα να ε, αναχαιτήσουμε τις αρνητικές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει όμως να θέσουμε λογικούς στόχους και να εφαρμόσουμε και την ανάλογη πολιτική. Χρειάζονται μέτρα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνώ. Θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε την υπέρτατη αυτή προτεραιότητα ότι το 30% ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο 2030. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να προβλέψουμε ακριβώς τέτοια μέτρα σύνεσης για να προβλεφθεί απαραίτητη προστασία. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Και τώρα ο συνάδελφος Ρόναη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες τραγικών γεγονότων. Καθημερινά βλέπουμε τις εικόνες από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Ένα δισεκατομμύριο ζώα ε, έχουν πεθάνει ε, στις πυρκαγιές αυτές. Ε, χάνεται η βιοπικιλότητα και η καταστροφή στην Αυστραλία. Έχει επιπτώσεις παντού, διότι ο καπνός εξαπλώνεται. Στη Νέα Ζηλανδία έχει μαυρίσει το χιόνι και επηρεάζεται η ατμόσφαιρά μας από τις πυρκαγιές αυτές όπου στον κόσμο και να γίνει κάτι, εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ θα νιώσουμε τις συνέπειες. Στην Αυστραλία και μόνο έχουμε εξαφάνιση ειδών. Είναι ευθύνη μας να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα της γης μας. Είναι αξία η βιοπικιλότητα. Ο Στεφανούτσα για ένα λεπτό. Eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi despre Ε, δεν θα μιλήσω για τα δάση σήμερα, θα μιλήσω για τις πόλεις. Το 60% του ανθρώπινου πληθυσμού το 2015 κατοικούσε σε πόλεις. Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή του κλίματος οδηγεί σε περισσότερους καύσονες ε, και, ε, θα, ε, και βλέπουμε και πιο ακραία φαινόμενα όσον αφορά τον Ιετό. Το Βουκουρέστι προσπαθεί με πράσινες περιοχές να λύσει τα προβλήματα αυτά και με πράσινες ταράτσες. Ε, μια έξυπνη πόλη σημαίνει βιώσιμη πόλη. Τα φυσικά οικοσυστήματα θα πρέπει να διατηρηθούν με σχετικούς διαδρόμους. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές επενδύσεις για κάτι τέτοιο πάρκα, ε, πράσινες προσώψεις κτηρίων, πράσινες ταράτσες μπορούν ε, να αποτελέσουν περισσότερες ε, πράσινες εκτάσεις για τους πολίτες μας. Η φύση δεν πρέπει απλά να είναι κάτι που σκεφτόμαστε στις διακοπές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ε, βλέπουμε τώρα την ε, έκτη καταστροφή ειδών που οφείλεται στον ε, άνθρωπο. Ένα εκατομμύριο ειδών απειλούνται. Οι στόχοι είναι καλοί, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να θέσει στόχους, για παράδειγμα, στην κοινή γεωργική πολιτική. Η γεωργία στην Ευρώπη συμβάλλει στην ε, εξαφάνιση ειδών. Θα πρέπει λοιπόν να διατυπώσουμε σαφείς στόχους για μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων ε, και ε, μείωση του αζότου. Εισάγουμε τεράστιες ποσότητες σόγιας, ενώ ταυτόχρονα επιδοτούμε την γεωργία στην Ευρώπη. Ο στόχος του 30% φαίνεται καλός, αλλά πρέπει ε, να έχουμε λιγότερο εντατική γεωργία και δασοκομεία. Έχουμε υποβάλει τροπολογία, ε, ένα μορατόριουμ για ε, την γενετική τεχνική, για, τις, για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταβίντ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν το δεν είναι συμβαλόμενο μέρος τη Συμφωνίας για την Διοπικιλότητα του ΟΗΕ. Συμβαλόμενα μέρη είναι τα κράτη-μέλη. Αυτό το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμα μία απόπειρα να χρησιμοποιήσει τα λεφτά των φορολογουμένων για διάφορα project για να υπερασπιστεί τη βιοπικιλότητα και να καταπολεμήσει υποτίθεται την ε, κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να συνάψει συμφωνίε όπω η συμφωνία με το Μερκοσούρ που καταστρέφει τροπικά δάση. Προκειμένου να εκτραφούν βοηθοί και να εξαχθούν ε, προϊόντα με βάση τη σόγια. Οι μεγάλες πολυεθνικές καταστρέφουν τη φύση και οδηγούν με τις δραστηριότητες τους σε υπερεκμετάλλευση. Υπάρχει επίσης μια αλληλευτική συμφωνία που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές, η οποία δεν βοηθάει τους γηγενείς πληθυσμούς. Αυτά κάνει στην πραγματικότητα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Κόκαλης. Για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Uh, uh, Σήμερα ψηφίσαμε συντεπτικά υπέρ της uh, ανακοίνωσης Κομισιόν ε, για την ε, Πράσινη Συμφωνία. Εκεί η Κομισιόν προτείνει να αναλύσουμε τα πορίσματα της, του IPPC για τους ωκεανούς και προτείνει μέτρα για το θαλάσσιο τομέα. Πριν από μία εβδομάδα, μία ε, έκθεση για την ατμόσφαιρα και την ατμοσφαιρική επιστήμη οι ωκεανοί τα τελευταία χρόνια ε, καταστρέφονται πολύ περισσότερο, κατά 450% ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ε, οι ωκεανοί όμως απορροφούν ε, ε, την επιπλέον θερμότητα και μπορούν να απορροφήσουν τη θερμότητα που παράγεται από 3,6 δισεκατομμύρια βόμβες χειροσύμας στο σημερινό μας ψήφασμα καλούμε την Κομισιόν να δώσει και μια μπλε διάσταση στην Πράσινη Συμφωνία. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια πραγματική μπλε ευρωπαϊκή συμφωνία. Είναι και η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Βίζικ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η προστασία τη ε, βιοποικιλότητα σημαίνει η προστασία των συνθήκων ζωή. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Εξαρτόμαστε από τη βιοποικιλότητα για να διονύσουμε το είδο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την έκτη μεγαλύτερη εξάλληψη ειδών την, προσκαλούμε, την προκαλούμε εμείς. Για να σώσουμε τη βιοπικιλότητα θα πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα και τα, τους διάφορους πληθυσμούς ειδών θα πρέπει να έχουμε μεγάλες ε, περιοχές όπου δεν δημιουργούμε κτίρια και κόβουμε δάση. Θέλουμε να αφήσουμε χώρο στη φύση, πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Χαίρομαι για το ψήφισμα προστασίας της βιοπικιλότητας που λαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη. Αλλά ίσως δεν αρκούν αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, ξεχνάμε ας πούμε και διάφορα πράγματα όπως τα πρωτογενή δάση της Ευρώπης που είναι οι πραγματικοί μας φύλακες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα γιατί ξέρετε η ζωή μας από αυτό. Ο κύριος Ανδρίου, για ένα λεπτό. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα εδώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία πριν από 40 χρόνια, ε, μέσα σε 40 χρόνια ε, έχει έχουν εξαφανιστεί ε, τουλάχιστον ε, έχουν εξαφανιστεί διάφορα είδη και έχουν χαθεί και μεγάλες δασικές εκτάσεις μέσα σε 10 μόλις χρόνια. Ε, έχουμε εμείς οργανώσει την υπερεκμετάλλευση των πόρων, οι κλιματικές αλλαγές και η ρήπανση. Εμείς είμαστε όλοι οι υπεύθυνοι για τις καθημερινές κακές μας συνήθειες. Είμαστε όμως και υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφή εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, συνάδελφοι, με κάποιες από τις αποφάσεις μας, όπως για παράδειγμα τις εμπορικές μας συμφωνίες με χώρες στην άλλη άκρη του κόσμου ή ε, με το άμεσο κέρδος που πριτανεύει σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος περιβάλλοντος ή των οικοσυστημάτων. Ε, εδώ λοιπόν, ε, εάν εμεί τα ανθρώπινα όντα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε λες και είμαστε το μόνο είδο επί του πλανήτη, θα καταλήξουμε να μείνουμε μόνοι μα. Γιατί θα έχουμε ε, προκαλέσει μόνοι μα την εξαφάνισή μα. Έχει φτάσει πια η στιγμή να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική εικόνα και αν δεν προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα θα πάψουμε να υπάρχουμε. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τώρα η κυρία Γιώβεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τα οικοσυστήματα και την προστασία των ειδών. Όλα αυτά, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και την προστασία των ειδών. Εδώ και χρόνια είμαστε μάρτυρες της ε, απώλειας, της εξαφάνισης πολλών ειδών, λόγω της εντατικής ε, γεωργίας, της χρήσης των φυτοφαρμάκων, της ρήπανση. Και τα αποτελέσματα είναι ότι η γη χάνει όλο και περισσότερο από το γενετικό της υλικό, τους φυσικούς της, τους της πόρους. Η βιοπικιλότητα είναι θεμέλιο της οικονομίας μας, της κοινωνίας μας. Η τελευταία μας προσπάθεια στρατηγική για τη βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει και πολλές ελπίδες. Όμως έχουμε ακόμη χρόνο για να κάνουμε κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τώρα να χαράξει μια επιτυχή στρατηγική να δώσει κάποιο ε, πρώτο δείγμα ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την νομοθεσία μας και την επικοινότητα. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Και τώρα ε, ο συνάδελφος Μέτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ δεν έχουμε μόνο κατεπήγουσες κλιματικές ε, κρίσεις να αντιμετωπίσουμε και συνέπειες, αλλά και σε σχέση με την επικοινότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι χάνουμε έντομα και ζωικά είδη είναι η έκτη μαζικότερη εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη και πρέπει να δούμε τι κόστο σημαίνει αυτό, τι τίμημα για τις μελλοντικέ γενναίες. Θα πρέπει να θα χρειαστούν μάλλον δεκαετίες για να αποκατασταθεί η βιοπικιλότητα, ενώ μέσα σε πολύ λίγο διάστημα μπορούμε να εξαφανίσουμε ε, ήδη το ένα μετά το άλλο. Είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Χρήση των φυτοφαρμάκων, ε, τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά, οι μονοκαλλιέργειες, όλα αυτά πρέπει να πάυσουν η προστασία της φύσης πρέπει να ε, επεκταθεί. Τα ύδατα, τα δάση, όλα τα οικοσυστήματα πρέπει να προστατεύονται. Χωρίς την προστασία και την ε, σωστή παραγωγή, η βιοπικιλότητα ε, δεν θα είναι το μόνο που θα φανιστεί, αλλά μαζί της και η ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε. Και τώρα, Γόλας, για ένα λεπτό. Παρακαλώ, Νίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πέρσι στην ε, ε, Παγκόσμια Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα αναφέρθηκε η μείωση των επικονιαστών και η απώλεια της βιοπικιλότητας. Το τμήμα αυτό της έκθεσης περιγράφει την πολιτική της Ιρλανδικής κυβέρνησης και <clears throat> το ότι γνωρίζει παντελώς την βιοπικιλότητα η κυβέρνηση της Ιρλανδίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραβεύει την εντατική γεωργία εις βάρος ε, της ε, φύσης. Και βλέπουμε εδώ παραβίαση των βασικών αρχών της βιοπικιλότητας. Χρειαζόμαστε νομικά δεσμευτικούς στόχους σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επαρκή χρηματοδότηση ε, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε επίσης ε, καλύτερη επιβολή το, της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την προστασία της φύσης. Πρέπει να ενηγήσουμε τώρα, αλλιώς θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μπούντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η βιοπικιλότητα αποτελεί μια από τις βασικές αξίες ε, της ανθρώπινης ζωής. Ε, από την άλλη, η βιοπικιλότητα ωφελεί όχι μόνο εμάς, αλλά και την επόμενη γενιά. Ο ανθρώπινος παράγοντας όμως έχει οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό της βιοπικιλότητας, ε, με σημαντικές επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα. Η αλλαγή του κλίματος είναι ιδιαίτερα πλευρή. Η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μέσο, μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν ε, ε, να ε, προστατεύσουν τη βιοπικιλότητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν ότι απαιτείται επαρκή χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η γεωργία θα πρέπει, ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να είναι εταίρος μας. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη γεωργία ώστε να προστατεύει καλύτερα το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Απαιτούνται έρευνες στην διατήρηση της βιοπικιλότητας και θα πρέπει αυτή να υποστηριχθεί με τους απαραίτητους πόρους. Ευχαριστώ, Βόντεν. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, η κυρία Βόντεν. Ε, δεν έχει σημασία που καθόμαστε στο Κοινοβούλιο ή που βάζουμε σταυρό στο ψηφοδέλτιο. Δεν παίζει ρόλο το χρώμα του δέρματός μας ή η γλώσσα που μιλάμε. Η βιοπικιλότητα που κληρονομήσαμε είναι πολύτιμος πόρος ε, που ε, ανήκει σε όλους μας και που θα πρέπει να προστατεύσουμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας οι καταστροφικές πυρκαγιές στην ε, Αυστραλία όπου ε, πιστεύετε ότι έχουν ε, πεθάνει ένα εκατομμύρια ζώα θα πρέπει να αποτελέσει ξυπνητήρι για όλους μας. Θα πρέπει να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους για να προστατεύσουμε την φύση και να μετριάσουμε την αλλαγή του κλίματος. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 δεν θα επιτευθούν. Ας κάνουμε καλύτερη δουλειά με τους στόχους του 2030. Ε, αύριο τελευταία φορά θα εγκαταλείψω το Κοινοβούλιο. Ε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, σας παρακαλώ να είσαστε προσιλωμένοι, να αντισταθείτε ε, στους πλούσιους, στα ε, συμφέροντα. Έναν πλανήτη έχουμε μόνο. Δεν θα είμαι εδώ για να ε, αγωνιστώ για τον πλανήτη αυτόν. Ε, εσείς όμως θα είσαστε εδώ. Σας παρακαλώ φροντίστε να αγωνιστείτε για τον πλανήτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο Σάλιβαν για ένα λεπτό. Παρακαλώ έχετε το λόγο η κυρία Οσάλιβαν. Η συνάντηση ΚΟΠ ε, στο, στην ε, Κίνα θα είναι σαν την ε, συνάντηση του Παρισιού, αλλά για τη βιοπικιλότητα. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει πόσο επίγει το θέμα του κλίματος. Καταλαβαίνουν όμως επίσης ότι το κλίμα και η κρίση της βιοπικιλότητας συνδέονται μεταξύ τους ως ε, παιδαγωγός και δασκάλα οικολογία, πάντα μου άρεσε να εξηγώ με παραδείγματα. Εάν δεν προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα θα φτάσει η ώρα που τα παιδιά δεν θα ε, μπορούν ε, να μαζεύουν άγρια λουλούδια και θα γνωρίζουν τις πεταλούδες και τις πασχαλίτσες μόνο από τα βιβλία. Ε, αυτή τώρα είναι η στιγμή για να σταματήσουμε να αναχαιτήσουμε την καταστροφή οικοσυστημάτων ε, και ειδών ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν ασχοληθούμε με το θέμα της γεωργίας και της αλίας. Σήμερα υπερψηφίσαμε ψήφισμα πάνω στην Πράσινη Συμφωνία που πιθανότατα είναι η πιο φιλόδοξη περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν γίνονται αρκετά όσον αφορά τον τρόπο που καλλιεργούμε και αλλιεύουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να ενεργήσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κάνευ για ένα λεπτό. Η προστασία και διατήρηση της βιοπικιλότητας δεν είναι μόνο ουσιαστική για την προστασία της, των φαρμάκων, της τροφής, αλλά και για την υγιή ζωή και τις βιώσιμες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει η βιοπικιλότητα και η προστασία του κλίματος να μπουν σε ένα πλαίσιο στα πλαίσια μιας ε, φιλοπεριβαλλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Η Κομισιόν θα πρέπει να εγγυηθεί ότι θα υλοποιηθούν οι στόχοι της ε, βιοπικιλότητα και να χρηματοδοτήσει βασικά project τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μου, τη Βουλγαρία, το... Ο μηχανισμός διασφάλισης του Natura 2000 δεν εφαρμόζεται λόγω των ανεπαρκών κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα των μεταφορών, πολιτική ε, προστασία των δασών, τουρισμού, ενέργεια κτλ. Ε, έχουμε αυτοκινητοδρόμους ε, πάρκα ε, που είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Θα πρέπει να έχουμε σωστά παραδείγματα για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να ελοπιθούν οι στόχοι της Ένωσης, να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα, Κάρλε Κίντ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πολύ έχουμε το μάτι στραμμένο στην Αυστραλία. Ας κοιτάξουμε από πιο κοντά κάτι που καίγεται εκτός από την Αυστραλία, τη γη της Αυστραλίας. Είναι η κορολογενής φράχη. Ε, με, την, ε, τα πλαστικά, τη μόλυνση, τις ε, δραστηριότητες, τα πετρέλαια κτλ. Πιο συνολικά, τα δύο τρίτα του θαλάσσιου περιβάλλοντος τροποποιήθηκαν ουσιαστικά από την ανθρώπινη δράση. Αλλά στο νερό περνάει λίγο απαρατήρητο αυτό. Ας έχουμε φιλόδοξους στόχους για να αποκαταστήσουμε την, το θαλάσσιο περιβάλλον. Ας είμαστε φιλόδοξοι για να προστατεύσουμε 100% τους ωκεανούς μας, οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δύο σημεία του ψηφίσματος είναι επίγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη ε, θαλάσσια περιοχή της Κόμινς, χάρη στις προτεραιότητές της, θα πρέπει όλα τα μέρη της σύμβασης να αναγνωρίσουν τον ωκεανό ως κοινό αγαθό της ανθρωπότητας, γιατί εξαρτάται τη ζωή μας. Ευχαριστώ. Και τώρα, Πάουλος, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έφερα μαζί μου κάτι. Μια έκθεση για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκόπηση και βεβαίως διατίθεται online σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Βλέπουμε ότι τελευταία πενταετία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Περιβάλλον δεν βλέπει πολύ καλά τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν είναι καλές οι συνθήκες και ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι όλα τα ζωικά και φυτικά είδη παγκοσμίω μειώνονται το δίδαγμα της έκθεσης αυτής είναι ότι επιτέλους κάτι πρέπει να κάνουμε για την βιοπικιλότητα και τα είδη, την προστασία των ειδών. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε διαχωρισμένα τις υπόλοιπε πολιτικές και να μην επενδύουμε όσα πρέπει. Δισεκατομμύρια επενδύονται σε άλλους τομείς και σε αυτό το πρόγραμμα, το Natura, δίνουμε κάτι λίγα ψίχουλα. Θα πρέπει λοιπόν με το ψήφισμα που έχουμε εγκρίνει σήμερα το πρωί να προχωρήσουμε και να βρούμε νέους τρόπους, να δούμε πώς η κοινή αγροτική πολιτική μπορεί να στηρίξει τους στόχους αυτούς. Ε, όλες μας οι πολιτικές ε, μακροπρόθεσμα να υποστηρίξουν την προστασία του περιβάλλοντος ε, και όχι μόνο στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο, ε, συνάδελφος Βάιντερ έχει ένα λεπτό. Ο, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρω ε, που γνωρίζουν πολύ καλά την ορνηθολογία. Ξέρουν εκατοντάδες είδη. Ε, και σπαράζει η καρδιά μου που δεν μπορεί να δει μαύρους περλαργούς πια και διάφορα άλλα είδη. Κάθε μέρα 150 είδη ε, από φυτά και ζώα και ζώα της θάλασσας καταστρέφονται λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητα. Θα πρέπει να μειώσουμε την εντατική γεωργία και τη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων και ζυζανιοκτώνων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη βιολογική γεωργία και τροφή χωρίς γενικά τροποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να βελτιώσουμε την υγεία των φυτών και ζώων. Επίσης, τα οργανικά βιολογικά προϊόντα είναι πιο υγιή και πιο νόστιμα. Επίσης, αυτό έχει και οικονομικά ωφέλη. Όταν θα αυξηθεί η παγκόσμια ζήτηση για καθαρά τρόφιμα. Θέλω να υπάρχει καθαρή στήριξη για την βιολογική γεωργία και την καλή χρηματοδότηση, τη σωστή χρηματοδότησή της από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Η ε, κυρία Ριβαζή, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και δέκα χρόνια η αντίληψή μας και κατανόηση για την ελεξάρτηση χλωρίδας πανίδας και ανθρωπότητας έχει προχωρήσει. Όμως η καταστροφή συνεχίζεται με μια κλίμακα και διαστάσεις ανίποτες. Ε, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο ήδη βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 19 από το Παγκόσμιο Φόρουμ των ε, Επιστημόνων θα απειληθούν με εξαφάνιση. Έχουμε περάσει σε μια περίοδο ε, κρίσιμη που θα καθορίσει το μέλλον. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την προστασία τη βιοπικιλότητα και για ένα παράγοντα από τον οποίο θα κρυθεί το μέλλον τη ανθρωπότητα. Και όταν μιλάω για το μέλλον τη ανθρωπότητα, να θυμόμαστε ότι η απώλεια τη βιοπικιλότητα επηρεάζει του αυτόχθονε λαού, του ηθαγενεί. Αλλά όχι μόνο. Έχει να κάνει και με την διαφύλαξη τη βιοπικιλότητα και τον ε, ζωτικό ρόλο που εκείνοι διαδραματίζουν. Επίση, η απώλεια τη επικοινότητα έχει να κάνει με την επιστηστική την κυριαρχία και ανεξαρτησία των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι και να φύγει ένα ηχηρό μήνυμα από το Κουνμίνγκ στην Κίνα το 2020. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση, να καθαρίσουμε του ωκεανού και να ευνοήσουμε μια ε, καθαρή ε, γεωργία χωρί ε, γαματαφόμικων και χωρί φυτοφάρμακα. Ευχαριστούμε κυρία μου. Σα παρακαλώ να μην επερβαίνετε το χρόνο σα δεν θέλω να κόβω μικρόφωνα. Αποφεύγω να το κάνω, αλλά μην με υποχρεώσετε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Άριμοντ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να μιλήσω για την απόλυτα βιοπακυλαφητών και να πω ότι τα στοιχεία είναι παλιά. Ε, εδώ έχουμε χάσει ένα σωρό ε, έντομα και είναι πολλές οι οικονομικές απώλειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, θα πρέπει να ε, δούμε την απώλεια των εντόμων μαζί και τις μέλισσες. Η απώλεια των ειδών, η βιοπικιλότητα, έχει και οικονομικές συνέπειες και θα πρέπει και για οικονομικούς λόγους να προστατευτεί το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις μονοκαλλιέργειες, τις εντατικές, την εντατική γεωργία και τα νοικοτινοειδή. Θα πρέπει η προστασία του περιβάλλοντος να ε, μην μείνει στην τωρινή συμφωνία μόνο, αλλά να δούμε και τα σημεία των μονοκαλλιεργειών και των ε, φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει οι οικογενειακές επιχειρήσεις να προστατευθούν, καθώς και οι μέλισσες ε, ή όλα τα, όλες οι καλλιέργειες, σε αντίθεση με τα νοικοτινοειδή, εάν εξαφανιστούν οι μέλισσες θα χαθεί και η ανθρωπότητα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος, η συνάδελφος Βίνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε Πρόεδρε, συνάδελφοι, έχουμε ακούσει πολλά για την βιοπικιλότητα. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σύντομο λεπτό που έχω στη διάθεσή μου να πω ότι η βιοπικιλότητα έχει να κάνει και με τα οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα που μολύνονται κυρίως στο επίπεδο των εδαφών. Έχουμε πάρα πολλά μικροβιολογικά, καθαρισμό του νερού, φιλτράρισμα ε, που λειτουργούν χάρη στο καθαρό έδαφος. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν και τα εδάφη και οι γέες διότι χωρίς ε, σωστό και υγιές έδαφος ε, όλα απειλούνται. Θα πρέπει ε, να μην να εμποδίσουμε τη διάβρωση, να εμποδίσουμε την καταστροφή των έδαφων και την ρήπανσή τους και να δούμε ότι οι δικές μας ασθένειες πολλές φορές οφείλονται στο ότι έχουν αρρωστήσει τα εδάφη. Είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα και αφορά όλη την διαβίωσή μας. Θα πρέπει λοιπόν να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για την προστασία ακριβώ των εδαφών και των γεών. Ευχαριστώ η κυρία Σπυράκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Συγκεβίτσιους, είναι προφανέ από τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι χρειαζόμαστε επιγόντω μια νέα δεσμευτική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα οι πυρκαγιές στον αρκτικό κύκλο στον αμαζόνιο στην αυστραλία επανέφεραν στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη να υιοθετήσουμε δεσμευτικούς στόχους για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. με αυτό το όπλο οφείλουμε να εμφανιστούμε στην cop δεκαπέντε στην κίνα με αυτό το όπλο οφείλουμε να θέσουμε όλες τις δυνάμεις του πλανήτη ενώπιον των ευθυνών τους και να ζητήσουμε μια συμφωνία δεσμευτική ανάλογη με αυτή του παρισιού προηγουμένω όμω οφείλουμε ω ευρωπαϊκή ένωση να αναλάβουμε τι ευθύνε μα με επαρκή χρηματοδότηση από τον νέο προπολογισμό με την προστασία τη βιοποικιλότητα με την υποστήριξη των καθαρών τροφίμων και των παραγωγών του αλλά και με την εμπλοκή των επιχειρήσεων. οι καλέ πρακτικέ για την προστασία τη βιοποικιλότητα από επιχειρήσει όπω είναι το business for nature που εφαρμόζεται και στην ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό μα. σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Και δίνει το λόγο στον κύριο Μπίχνερ. Ένα λεπτό. Πολλά είδη ζώων, φυτών και άλλων οργανισμών λόγω της τεράστιας χρήσης χημικών θα εξαφανιστούν. Αλλά και επειδή εμείς ε, κατακτάμε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου όπου ζουν. Πολλά είδη πεθαίνουν χωρίς να τα παίρνουμε καν χαμπάρι από την ακτινοβολία η οποία αυξάνεται όλο και περισσότερο. Μακροχρόνια έρευνα έχει δείξει ότι η ακτινοβολία για παράδειγμα στις μέλισσες και σε άλλα ζώα προκαλεί απώλεια του προσανατολισμού, της αίσθησης προσανατολισμού. Οπότε φεύγουν από εκεί που κατοικούν αλλά δεν μπορούν να ξαναβρούν το σπίτι τους. Τα ποντίκια μερικές φορές ε, στην πέμπτη γενιά ε, γίνονται, ε, χάνουν την δυνατότητα να αγωνιμοποιήσουν. Εάν συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την κινητή τηλεφωνία, πολλά είδη φυτών και ζώων θα εξαφανιστούν ε, ανεπιστρεπτοί από αυτή τη γη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για τη στρατηγική μα, διότι είναι και θέμα τι γίνεται με τι θάλασσε. τι γίνεται με του ωκεανού που απορροφούν πάνω από 25% των ε, βλαπτικών εκπομπών. Είναι ο πιο μεγάλο μας πάροχος του, του, ε, του οξυγόνου και γι' αυτό και με τη συμφωνία του Παρισιού είπαμε ότι έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αθεκτικοί, να προσαρμοστούμε στα τις αλλαγές του κλίματος, Οπότε έτσι να μπορέσουμε να μειώσουμε το οξυγόνο, εκείνο το οποίο δεσμεύουν οι ωκεανοί, 14% με το 2050. Αυτό όμω θα είναι πάρα πολύ κακό για τους βιώτοπους και για ό,τι έχει σχέση με του ωκεανούς. Έχουμε ένα δις ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και επίση ε, έχουμε αύξηση του πλαστικού 17 φορές ε, πιο μεγάλο συνόγκο των πλαστικών από την Πορτογαλία. Και επομένω οι ωκεανοί θα πρέπει να διασωθούν και έτσι να κερδίσουμε τη μάχη της βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για τον κύριο ε, Λίζα του δώσω ένα λεπτό γιατί θα αργήσει να έρθει. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε παγκοσμίω και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την προστασία των ειδών. Γι' αυτό θα ε, ψηφίσουμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος ως ΕΛΚ αύριο και ευχαριστώ ε, κυρίως την Αγνές Ευρέν εκ μέρους του ΕΛΚ. Θέλω να προειδοποιήσω ότι όταν μιλάμε για βιοποικιλότητα πάμε πάντα και ψάχνουμε την απλή λύση, περισσότερη προστασία των χώρων, ε, αυστηρότερες ποινές ε, για παραβίαση συνθήκων. Να βρούμε και νέες ιδέες, καλύτερη δικτύωση και όπως πρότεινε ο συνάδελφος Γιάρα στη μεταρρυθμίση της γεωργικής πολιτικής ε, καλύτερη άρδευση κάποιων καλλιεργήσιμων χώρων. Μερικές φορές όταν Ε, η προστασία ε, της φύσης έρχεται σε αντίθεση με κάποια προβλήματα, με θέματα υγείας. Δεν πρέπει να κατηγορούμε μόνο τη γεωργία μόνο μονομερός. Αυτό δεν μας οδηγεί προς το στόχο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και όχι ο ένας εναντίον του άλλου. Ευχαριστώ πολύ. τώρα αρχίζει το Τρει έχουν ζητήσει τον ε, λόγο και οι τρει θα καλυφθούν και ξεκινούμε από τον κύριο Νόβακ. Την κυρία Νόβακ. Είναι σαφές ότι θα υποφέρουμε και αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζωικά είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι όμως και ρεαλιστικά. Οπότε οι πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν για τα διοικητικά μέτρα. Κάθε ζωικό είδος έχει τη δικιά του λειτουργία και πρέπει να το επιτρέψουμε να τη φέρει σε πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Πώς να προστατεύσουμε όλα τα είδη του ζωικού και του φυτικού βασιλείου, αλλά συγχρόνως να ικανοποιήσουμε και τις ε, ανάγκες των ανθρώπων. Δεν φταίνουν οι αγρότες για όλα αυτά. Και οι καταναλωτές έχουν τις δικές τους ευθύνες και πρέπει να τις αναλάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νόβακ, ο κύριος Χάισελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πράγματι η ζωή στον πλανήτη αυτό απειλείται και δεν πρόκειται μόνο για την κλιματική αλλαγή, πρόκειται και για την μείωση της βιοπικιλότητας. Και το βλέπουμε αυτό, αυτές τις απειλές, όχι μόνο με τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο που κάηκε, αλλά και στη Σιβηρία Επίσης βλέπουμε ότι μειώνεται ο αριθμός των μελισσών. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς θεωρούσαμε ότι αποτελούν κομμάτι της ζωής μας όταν πηγαίναμε βόλτα στη φύση. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα νοικοτοειδήτα επικίνδυνα, δηλαδή φυτοφάρμακα, να πάψουμε να κόβουμε τα δέντρα. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε αυτή τη συζήτηση και που θα ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα αύριο. Πρέπει οι χώρες μέλη να κάνουν περισσότερες προσπάθειες και να δοθούν αρκετά χρήματα ώστε τα μέτρα να είναι δεσμευτικά. Να βρούμε χρήματα από το προπολογισμό αλλά και από άλλα οριζόντια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χάισελ. Ακολουθεί συνάδελφος Φερέρα. Ευχαριστώ. Στόχος μας είναι να μειωθεί η απώλεια της ε, βιοπικιλότητας. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέρνουμε. Τα διάφορα είδη, ζωικά και φυτικά, μειώνονται. Κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Με πολύ σημαντικέ συνέπειες για το ανθρώπινο είδος. Εδώ δεν φτάνει να παριθμούμε στρατηγικές που έχουν αποτύχει μέχρι τώρα ή να βάζουμε φιλόδοξους στόχου, Χρειάζονται φιλόδοξα μέσα. Στα πλαίσια λοιπόν του επόμενου προγράμματος CFP θα έλεγα ότι ούτε και εκεί τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχουμε καταλήξει να εμπορευόμαστε τη φύση και τους σπόρους της. Αυτό όμως επιδεινώνει την κατάσταση. Η καταστροφή των οικοτόπων, ε, η εισαγωγή ειδών, τα οποία όμως ε, σκοτώνουν άλλα. Είναι ένα οικονομικό μοντέλο που δεν είναι καλό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε, τις ρίζες του κακού και να αμφισβητήσουμε ακριβώς αυτό το μοντέλο και αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστούμε κύριε Φερέρα. Κλείνει, έκλεισε τώρα το κατσιάι Και τελευταίος θα μιλήσει ο κύριος Επίτριο Πώς Σίνκεβίτσιος. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ομιλίες σας και για την υποστήριξή σας για μια φιλόδοξη πολιτική βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Λένα που είπε ότι δεν έχουμε παρά έναν πλανήτη. Δεν υπάρχει δεύτερος. Έχουμε τεράστια ευθύνη να υλοποιήσουμε το μετασχηματισμό που χρειάζεται για να επιστρέψει μέχρι το 2030 στην ανάκτησή της η φύση, να αποκατασταθεί η φύση προς όφελο όλων των ανθρώπων. Πρέπει να είμαστε πράγματι φιλόδοξοι, πρέπει να εξηγήσουμε καθαρά στους πολίτες και στους ενδιαφορομένους για ποιο λόγο χρειάζεται να αλλάξουμε τους τρόπους κατανάλωσης και παραγωγής, να επισημάνουμε τα ωφέλη της ευημερία, της υγείας ε, και να διασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση για την οικονομία. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι έχω σημειώσει επαρκώς και άκουσα προσεκτικά τις εκκλήσεις σας ε, για δεσμευτικούς νομικά στόχους. Τα σχόλια σας για τα, τη ζενιοκτώνα, τη γεωργία, την αποδάσωση ε, και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εξακολουθούμε να συζητάμε εσωτερικά την στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, αλλά οι στόχοι που θα προσανατολίζονται σε δράση θα πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους τομείς πολιτικής συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκομείας και της αλληλεία. Και όσον αφορά την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης. Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και να έχουν αξιολογηθεί επαρκώς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Σάλιβαν, τον κύριο Μέλλο, τον κύριο Καλασκίνη, επειδή επισήμαναν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι ωκεανοί, όχι μόνο για τη βιοπικιλότητα, αλλά και για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ως Επιτροπός για το Περιβάλλον, τους ωκεανούς και την Αλία, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο